και την τεχνολογία σε τρίτες χώρες. Έχει τον λόγο η συγγήτρια παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και τελικά η τεχνολογία μας βοηθά. Κύριε Αντιπρόεδρε Τίμερμαντς, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί σκιώδεις συγγητές, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, συνεργασία που είχαμε για την έκθεση αυτή και να ευχαριστήσω και όλα τα άτομα αυτά παγκοσμίω, τα οποία κατάφεραν μέσω διαδικτύου να μου στείλουν πάρα πολλέ νοθεσίε και προτάσει και κατά αυτόν τον τρόπο η έκθεση που ψηφίσαμε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων που θα ψηφίσουμε αύριο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γίνεται πιο ισχυρή. Το crowdsourcing λοιπόν λειτουργεί. Ξέρετε ότι η τεχνολογία πραγματικά προωθεί αλλά μπορεί και να περιορίσει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η τεχνολογία μπορεί να μα βοηθήσει να έχουμε καλύτερη πρόσβαση στην ελεύθερη έκβραση καθώ επίση και στο δικαίωμα του συνέχερστε αλλά την άλλη όμως μέσω της τεχνολογίας μπορούμε να έχουμε ακόμα και κάποια φαινόμενα διαφθοράς, αλλά μπορούμε και να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά. Η παρακολούθηση των εκλογών, η αντιμετώπιση φυσικών καταστραφών, όλο και περισσότερο μπορεί να διευκολυνθεί μέσω της τεχνολογίας. Τα τεχνολογικά όμως συστήματα μπορεί και να τύχουν κατάχρηση, μπορούν να αποτελέσουν εργαλεία για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω της μαζικής παρακολούθησης ορισμένων ανθρώπων, μέσω της παρίσφρησης, της παρακολούθησης, της κατασκοπίας. Πέρα λοιπόν από τις τεχνικές προδιαγραφές, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ακριβώς πώς χρησιμοποιούνται τα συστήματα πληροφορικής και αν τελικά τα εργαλεία πληροφορικής προωθούν ή καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ποια αρχή, ποιος χρήστης, ποιος παρακολουθεί τη σωστή χρησιμοποίηση αυτών των μέσων. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να δούμε όλε αυτέ τι πλευρέ και θα πρέπει να τι αξιολογήσουμε στα πλαίσια τη ευρωπαϊκή πολιτική. Μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία απαιτείται, ιδίω για τι τεχνολογίε εκείνε οι οποίε προωθούν την παρίσφρηση και την παρακολούθηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και νομίζω ότι εδώ πολλέ φορέ δημιουργείται μία λανθασμένη διάκριση ανάμεσα στην ελευθερία και την ασφάλεια ή το, γεγονό ότι πολλέ φορέ η προώθηση τη ασφάλεια χρησιμοποιείται ω πρόσχημα για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προώθηση τη ασφάλεια και προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει από κοινού να προωθούνται, τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρί να έχουμε παράλληλα πολιτικέ οι οποίε βάλουν κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εδώ πέρα στα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και στα πλαίσια συγκεκριμένα τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση βλέπουμε ότι πολύ συχνά δεν μπορούμε καν να προστατεύσουμε του ίδιου εργαζόμενού μα, του ίδιου του διπλωμάτε μα από τα συστήματα αυτά τα οποία συζητάμε σήμερα. Στι συστήματα πληροφορικής μυστικών πληροφοριών hackers πολλές φορές χρησιμοποιούν παρισφρετικές τεχνολογίες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί εδώ στην Ευρώπη και η αξιοπιστία της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπονομεύεται άμεσα όταν μια Ιταλική εταιρεία άδικα έχει το δικαίωμα να πουλήσει τεχνολογίες πληροφορικής στο Σουδάν ή σε άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν κάτι τέτοιο συμβαίνει με κάποια γαλλική επιχείρηση ακόμα και αν νομίζουμε τελικά ότι η παροχή αυτή τεχνολογιών προστατεύεται από κρυπτογράφηση. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί περασπιστέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν, στη Ρωσία, σε πάρα πολλέ χώρε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση που θα πρέπει με τι τεχνολογίε τη πληροφορική Ευρωπαϊκή Ένωση να προστατεύονται και όχι να υπονομεύεται. Η πολιτική λοιπόν τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενσωματώνει τη διάσταση τη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στι τεχνολογίε που χρησιμοποιούμε και θα πρέπει αυτό να διέπει όλε τι πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείτε να βρείτε πολύ συγκεκριμένε προτάσει στην έκθεση αυτή. Λέμε συγκεκριμένε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να απαγορεύονται οι μηχανισμοί κρυπτογράφηση, ή σε καμία περίπτωση θα πρέπει να δίνονται τα password όσον αφορά αυτέ ε, ε, ε, τι πολιτικέ τα μέσα κρυπτογράφηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προστατεύσουμε πληροφοριοδότες ή υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υπερασπιστε ανθρωπινων δικαιωματων εκτο ευρωπαικη ενωση η ευρωπαικη ενωση θα πρέπει να γίνει παγκόσμιο ηγέτη και να καταφέρνει να διασφαλίσει ότι όντω η τεχνολογία προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν δώσουμε εμεί το θετικό παράδειγμα. Ευχαριστώ. Ε, σα ευχαριστούμε. Περνάμε στη διαδικασία Catch the Eye και σα ενημερώνω ότι θα ακούσουμε πέντε ομιλητέ σε Catch the Eye για κάθε έκθεση για να μοιράσουμε δίκαια το χρόνο. Κύριε Πόλσακ, ένα λεπτό και θέλω να τονίσω ότι όσοι μίλησαν ε, σε προηγούμενες συζητήσεις ε, ίσως ε, να μην επιλεγούν για το Catch σε επόμενες συζητήσεις. Θα προσπαθήσω να είμαι δίκαιη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για αυτή την τόσο σημαντική έκθεση. Πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα εύστοχο το περιεχόμενό της. Το ζήτημα που πρέπει να μας απασχολεί είναι ποια τιμή, ε, πόσο τιμάται η συνείδησή μας ε, και πόσο θα πουλήσουν τη δική του συνείδηση οι επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις ε, που θα ήταν αδιανόητες όχι μόνο για την τσεχική δημοκρατία αλλά και γενικότερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ζήτημα της έκθεσης είναι σε ποιο βαθμό μπορούν να μεταφερθούν στοιχεία που σχετίζονται με βασικά ανθρώπινα δικαιώματα σε τρίτες χώρες. Εγώ Πιστεύω ότι υπάρχουν οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα που οφείλουμε να προστατεύουμε. Πρόκειται για μια αξία που ε, υπερβαίνει αυτή της απασχόλησης ε, ή του ΑΕΠ. Δυστυχώς δεν μοιράζονται όλοι αυτή την άποψη και θα πρέπει να βρούμε ένα ε, σύνορο και μια κόκκινη γραμμή. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Καπούτο τώρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Βλέπουμε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προκύπτουν από χρήση νέων τεχνολογιών, ε, κυρίως στο διαδίκτυο. Οι παραβιάσεις ε, σχετίζονται με δικαιώματα και ε, κώδικες διοντολογίες που σχετίζονται με την χρήση των νέων τεχνολογιών ε, με στόχο την παρακολούθηση ή την παρίσχρηση. Ex-post έλεγχη είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Παρότι υπάρχει ευγενής χρήση των νέων τεχνολογιών, ε, θα πρέπει να προσέξουμε ε, και να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των πλέον ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων. Θα πρέπει λοιπόν ε, ιδιαιτέρως να προσέξουμε ό,τι σχετίζεται με τις έρευνες, την παρακολούθηση και ούτω καθεξής. Όλοι θα πρέπει δεν να εμπλακούν σε αυτούς εξ post ελέγχους. Ευχαριστούμε κύριο Τζάκους για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να συγχαρώ την ναι, κυρία Σάκα για αυτή την έκθεση. Θα ήθελα να πω ευθύς εξ αρχής ότι το διαδίκτυο έχει διανοίξει πολύ σημαντικούς νέους τομείς ελευθερίας. Ωστόσο αυτό μου θυμίζει τον Άλφερντ Νόμπελ που εφήβε τον ε, δυναμίτη, την νητρογλυκερίνη και ε, με την ε, επινόησή του, με την εφεύρεσή του αυτή ε, διανοίχτηκαν άπειρες νέες δυνατότητες. Ωστόσο πρέπει να δούμε ότι υπάρχουν και δυνατότητες κατάχρησης που διανοίγονται από δικτατορικά καθεστώτα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρκετά κερδοφόρες συμφωνίες και είναι σημαντικό το ότι αυτή η έκθεση πρέπει ε, να μας κάνει να λάβουμε υπόψη οποιασδήποτε δυνατότητες κατάχρησης στο μέλλον και να λάβει υπόψη η Επιτροπή αυτό το στοιχείο. Χάουταλα παρακαλώ στη συνέχεια. Ευχαριστώ Πρόεδρε, Αντιπρόεδρε της Επιτροπής. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις από τις τεχνολογίες αυτές ε, στα δικαιώματα του ανθρώπου για τις γνώσεις, ε, για τα στοιχεία, για τα δικαιώματα του ανθρώπου, αλλά υπάρχει και παγίδα εδώ όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και η κυρία Σάκες συνέταξε μια εξαιρετική έκθεση και πρέπει να αναγνωρίσουμε νομίζω ότι η Ευρώπη, οι επιχειρήσεις της Ευρώπης, το γεγονός ότι υπάρχει υπονόμευση της αξιοπιστίας μας όσον αφορά τις παραβιάσεις δικαιωμάτων του ανθρώπου στο Ιράν, στο Ουσμπεκιστάν, σε πολλές άλλες χώρες και με τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας. Πρέπει επίσης εδώ να αναφέρουμε ότι αυτό που αναφέρει η έκθεση ότι οι υπηρεσίες και το δίκτυο, τα δίκτυα θα πρέπει να μπορούν να ε, φωτίσουν τα δίκτυα τα οποία μπορούν να δημιουργηθούν και τις δυνατότητες για καταπιεστικά καθεστώτα. Υπάρχουν πολλά καλά στοιχεία σε αυτή την έκθεση και πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί να αποφύγουμε περί τη λογοκρισία στο διαδίκτυο ιδίως παρότι πιστεύω ότι αυτό επιτυγχάνεται καλύτερα από τις εθνικές κυβερνήσεις και όχι από τελεσίγραφα και κελεύσματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το εδάφιο 17 της έκθεσης, δηλαδή όσον αφορά το εμπόριο και την επιβολή των δυτικών αξιών σε τρίτες χώρες ως όρο για την ανάπτυξη του εμπορίου με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Για μένα αυτό δεν είναι μόνο απαράδεκτο, αλλά είναι το άκρο ναότον της αλαζονίας. Ε, δεν είναι δυνατόν εμείς να γνωρίζουμε καλύτερα και να λέμε τι θα έπρεπε εκείνες να κάνουν. Και πραγματικά αυτό περιφρονεί τη δική, τα δικά του κυριαρχικά δικαιώματα. Δεν μπορώ λοιπόν να υποστηρίξω μια έκθεση που συμπεριλαμβάνει τέτοιου είδου διατυπώσει. Ο κύριος Τίμεμας θα λάβει τον λόγο για να απαντήσει στα θέματα της συζήτησης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Σάτια για την πολύ καλή αυτή έκθεση ε, και ορισμένες φορές ε, διαβάζουμε δημοσιεύματα για την αρνητική πλευρά των ε, νέων τεχνολογιών. Βλέπουμε πολυάριθμα εύστοχα σχόλια και ε, ιδέες ε, και μεγάλες προκλήσεις ε, για το μέλλον μέσα στην έκθεση. Φυσικά θέλουμε να τατικοποιήσουμε τις προσπάθειές μας ούτως ώστε να έχουμε μια δικαιότερη διακυβέρνηση στο διαδίκτυο αλλά να εξασφαλίσουμε και την ασφάλεια των δικτύων. Το ίδιο βλέπετε και στην πρόσφατη ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει τη δέσμευση σε όλου του τομεί εξωτερική δράση να προωθήσει αυτά τα δικαιώματα που σχετίζονται με τι νέε τεχνολογίε. Δεδομένη τη σημασία των νέων τεχνολογιών στην καθημερινή μα ζωή, με την πρόσβαση στην κινητή τηλεφωνία, στο ίντερνετ μάλλον, ε, ε, μέσω, των κινητών ε, μέσω της κινητής τηλεφωνίας και η σχέση που υπάρχει με τα ανθρώπινα δικαιώματα μας αναγκάζει να αντιμετωπίσουμε, να δείξουμε αυτό το θέμα σε προτεραιότητα. Είναι ρόλος κλειδί αυτό των ε, ε, ψηφιακών δικαιωμάτων ε, για να προστατεύσουμε και βασικές ανθρώπινες ελευθερίες. Βλέπουμε στην έκθεση, παραδείγματο χάρη υπάρχει το δικαίωμα στην έκφραση, στην ενημέρωση, στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών δεδομένων. Εκεί σημειώνονται παραβιάσεις λόγω της λογοκρισίας, της παράνομης παρακολούθησης, επαρίσφυσης, συλλογής ε, και διατήρησης ατομικών δεδομένων ε, που γίνονται σε μεγάλη κλίμακα για έκνομους ε, λόγους. Βλέπουμε λοιπόν ότι θα πρέπει οι να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε αυτά τα βασικά δικαιώματα και να προωθήσουμε τις δυνατότητες που έχουμε για δημοκρατικό έλεγχο, ούτω ώστε από οι αρχές επιβολής νόμου και δικαστικές αρχές να μπορέσουν να προωθήσουν την υπόπτη αυτών των δραστηριοτήτων εξασφαλίζοντας την ελευθερία ε, έκφρασης ε, ε, επιγραμμικά και μη. Θα προωθήσουμε λοιπόν αυτέ τι κατευθυντήριες γραμμέ, ακόμη και στι σχέσει μα με τρίτε χώρε αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει και καλωσορίζει την, το διορισμό ενό ειδικού εκπροσώπου του ΟΗΕ για τα δικαιώματα το δικαίωμα της ιδιωτικής ε, ζωής. Ε, βλέπουμε ότι η ανταπόκριση μας ε, στις τρομοκρατικές ενέργειες δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να πλήττει τα δικαιώματά μας, το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και τα ατομικά δεδομένα. Η ψηφιακή ατζέντα που δημοσίευσε φέτος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκαθάρισε ότι θα αλληληφθούν τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να υπάρξει συμμόρφωση, ασφάλεια και εξασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα των μέτρων που αναλαμβάνει. Θέλουμε να σταθούμε στο πλευρό των των προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ακτιβιστών τη κοινωνία των πολιτών και των εξαρτήτων δημοσιογράφων, ώστε να ε, χρησιμοποιήσουμε τι νέε τεχνολογίε για να αγωνιστούμε για την ελευθερία. Επίση, ε, η πολυφωνία των ΜΜΕ είναι και για μα προτεραιότητα και έχουμε δει ανεξάρτητα προγράμματα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μέσων Μαζική Ενημέρωση ε, και Τύπου ε, με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έτσι θα αντιμετωπίσουμε τι παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σχέση με τρίτε χώρε, ε, και θα προωθήσουμε τι δράσει. Ε, τα, συνοδεύοντας τις δράσεις μας με ψηφιακή ε, εκπαίδευση. Επίσης, ε, θα χρησιμοποιήσουμε κυρώσεις κατά των πολιταρχικών καθεστών που περιορίζουν αυτές, αυτά τα δικαιώματα Όπω στη Συρία παραδείγματο χάρη για τι εξαγωγέ ε, ε τις άδειες εξαγωγών ε, αναθεωρούμε την ε, δράση μας ούτω ώστε να μην χρησιμοποιούνται για παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το 2014 έχουμε εισαγαγεί νέου περιορισμού περιορισμούς εξαγωγέ εξαγωγές λογισμικού ε, και λογισμικών παρακολούθηση. και επίσης διερευνούμε περαιτέρω τι δυνατότητε που υπάρχουν να επεκτείνουμε ε, τους ελέγχους εξαγωγών, ούτως ώστε να χρησιμοποιήσουμε τις δράσεις μας και για τις παρακολουθήσεις ε, που γίνονται στο ε, κυβερνοχώρο και χρησιμοποιούνται για περιορισμό των ανθρωπίνων δικαιωματών. Όπως μας λέει η κυρία Σάτια μέσα στην έκθεσή της, όντω θα πρέπει να αντιληφθούμε ποιες είναι οι συνέπειες της χρήσης των νέων τεχνολογιών επί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις εξωτερικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεργαζόμαστε λοιπόν με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για να εξυπηρετήσουμε αυτό το στόχο στόχο οι τεχνολογίε χρησιμοποιούνται για να προωθήσουν ελευθερία σε παγκόσμιο επίπεδο και να, ε, τα, οι ωφέλειε που μπορούμε να αποκομίσουμε είναι μια κοινή ευθύνη για όλου, ε, για τον ιδιωτικό τομέα, για την κοινωνία των πολιτών, για τι κυβερνήσει, ε, για, τη, για του πολίτε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρόθυμη να επαναλάβει τη δέσμευση που έχει αναλάβει σε σχέση με την ελεύθερη πρόσβαση στι νέε τεχνολογίε χωρί διακρίσει, χωρί λογοκρισία. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Λίγη συζήτηση και θα ψηφίσουμε αύριο για αυτή την